κόλλησης της εφαρμογής των νόμων σε ευρωπαϊκό νόμο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Δαμανάκη. Κλείνει η συζήτηση. Η συμφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα την ερώτηση προς την Επιτροπή για την Συμφωνία τη Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας. Η κυρία Φράγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρωτόκολλο αλληλείας με τη Μαυριτανία εκπνέει στις 31 Ιουλίου του 2012 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Συμβούλιο εντονή για έναρξη των νέων διαπραγματεύσεων. Εξ όσων γνωρίζουμε, η πρόταση εντολής ήδη συζητάται από το Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει προσεχώς από πλευρά μα λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 218 της συνθήκης που ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει καθήκοντα για τις ε, τελικές συμφωνίες αλίας. Έχουμε ήδη εκφράσει την ε, πρόθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες που μας δίνονται τόσο από τη συνθήκη όσο και από την ε, διαθεσμική συμφωνία πλαίσιο για την συμμετοχή μας στις αλλιευτικές συμφωνίες και την πλήρη ενημέρωση και σε ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο θεωρούμε ότι πρέπει να δεσμευτούμε με, την ίδια διαδικασία, με τη διαδικασία αυτή ήδη από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό και η Επιτροπή Αλία αποφάσισε να ξεκινήσει με τη Μαυριτανία αυτή τη νέα διαδικασία, η οποία αφορά την παρουσίαση μια προφορική ερώτηση που θα μα δώσει τι πρώτε πληροφορίε για τη μελλοντική διαπραγμάτευση και την προετοιμασία μια πρόταση ψηφίσματο που θα περιλαμβάνει τι ανησυχίε μα για όλε τι συμφωνίε, σε αυτή την περίπτωση για τη συμφωνία με τη Μαυριτανία, ζητώντας να ληφθούν υπόψη από τους διαπραγματευτές και να συμπεριληφθούν στο τελικό πρωτόκολλο η συμφωνία με τη Μαυριτανία είναι ζωτική σημασία και για την ίδια τη χώρα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη Μαυριτανία σημαίνει το 29% συνεισφορά στον εθνικό προπολογισμό τη. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για μία από τι τρει κοινέ ε, συμφωνίε που επιτρέπουν ε, να υπάρχουν συγκεκριμένε ε, ρυθμίσει για την αλληλεία σε περιοχέ οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση η συμφωνία αυτής της μορφής και τα όσα γνωρίζουμε μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε συγκεκριμένες συστάσεις οι οποίες ε, θα συμπεριληφθούν στη συμβιβαστική πρόταση που θα συζητήσουν οι πολιτικές ομάδες τις επόμενες ε, εβδομάδες για να αναφέρουμε και κάποιες ανησυχίες που προκύπτουν από το πρωτόκολλο το οποίο ενισχύει και σε γενικές γραμμές είναι οι εξής. Καταρχάς, τη σημασία που προσδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, την, ε, για το χρηματοοικονομικό αντιστάθμισμα και τη σωστή του εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες του τομέα αλλά και ε, η αλλιευτική διοίκηση της Μαυριτανίας για να υπάρχει μια βιώσιμη πολιτική αλίας. Δεύτερον, ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η Κοινή Επιστημονική Επιτροπή και ε, τη σημασία του και την καλή του λειτουργία. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι πόροι για να μπορεί να δίνονται συστάσεις για τη βιολογική κατάσταση των ηχθειοαποθεμάτων καθώς επίσης και των ε, δυνατοτήτων που δίνονται ε, στους ε, αλλιευτικούς στόλους που αλλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και τι αλλιεύματα ε, έχουν τρίτες χώρες που αλλιεύουν στην περιοχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα μπορέσουμε να γνωρίζουμε ποια είναι τα ποσοστά αλλιεύματα που μπορεί να παραχωρήσει πραγματικά η Μαυριτανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης και την ανησυχία μας διότι αλληλευτικές συμφωνίες που θα διαπραγματευτούμε θα πρέπει ε, να είναι ρεαλιστικές και να μην ε, ε, πληρώνουμε παραπάνω από όσα θα έπρεπε. Πέραν από τις αλληλευτικές δυνατότητες θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση και για τα τεχνικά μέσα και μέτρα για κάθε είδος ώστε να μην καταβάλλονται κονδύλια για είδη τα οποία από τεχνικής πλευράς θα είναι πολύ δύσκολο ή έως και αδύνατο να αλλιεύσουμε. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε τι χρήση κάνει η Μαυριτανία των κεφαλαίων ελέγχου που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο, τόσο όσον αφορά στην ε, προτίμησή τους σε εναλλακτικές μεθέδους από το σε σχέση με το UVS, καθώς επίσης, VMS, ε, συγγνώμη, καθώς επίσης και το τι γίνεται με τις εκτιμήσεις. Είναι πολύ σημαντικό και οι δύο πλευρές να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί και θα πρέπει να συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνονται αυτές οι δεσμεύτες ε, στο μελλοντικό πρωτόκολλο. Κυρία Επίτροπε, θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, διαπραγματευτή να λάβει υπόψη και αυτές τις ανησυχίες και τα όσα θα περιλαμβάνονται στο ψήφισμα το οποίο θα υιοθετηθεί στην επόμενη Ολομέλεια και ήδη σας ανακοινώμενο ότι θα παρακολουθήσουμε επισταμένα το θέμα από πλευράς Επιτροπής Αλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φράγα, πρόεδρο της Επιτροπής Αλληλείας, για την προφορική αυτή ερώτηση. Πραγματικά είναι ιδιαίτερος ευπρόσδεκτη η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία. Εν γέννη συμμερίζομαι τις ανησυχίες της και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα είναι τα καλύτερα δυνατά. Θέλω να σας πω δύο λόγια για την ισχύουσα αλληλευτική συμφωνία με τη Μαυριτανία η οποία σκοπό έχει να διατηρήσει ε, και να εκμεταλλευτεί με βιώσιμο τρόπο τα αλληλευτικά αποθέματα, να καταπολεμήσει την παράνομη αλληλεία να προωθήσει την ανάπτυξη λιμενικής υποδομής και να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον. Μέσω, με αυτή τη συμφωνία έχουν περιοριστεί οι δυνατότητες αλίες και οι έχουν, μειωθεί, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι άδειε αλληλεία, ανατόνο και οι ποσοστώσει. Παρά τα αυτά, πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε το θέμα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συμφωνώ ε, επ' αυτού με την κυρία Φράγα. Η συμφωνία με τη Μαυριτανία έχει καταστεί η πιο σημαντική από χρηματοοικονομική πλευρά. Είναι ε, άποψη, είναι η πιο σημαντική από τη συμφωνία μας. Δεδομένης αυτής της εξέλιξης, η Κομισιόν μελετά την εισαγωγή ενός ε, σημαντικού στοιχείου αιρεσιμότητας σε σχέση με το πρωτόκολλο. Και αυτό, μεταξύ άλλων, μπορεί να γίνει με την με τη σύνδεση, με, την αποσύνδεση μάλλον της, των τιμών με την στήριξη του κλάδου. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ε, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και άρα να μην διαταραχθούν οι αλληλευτικές δραστηριότητες των ε, αλληλευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο ρυθμός εκτέλεσης της συμφωνίας ήταν πολύ ψηλός το 8 και το 9. Αντίθετα, το 2010 είχαμε πολύ χαμηλό επίπεδο ε, των κεφαλαίων, μόνο, 50% και αυτό λόγω του υψηλού ποσοστού παρακράτησης των ε, πόρων αυτών από τα Υπουργεία της Βρετανίας. Πέρυσι η συμφωνία με την μαυρετανική πλευρά αποφάσισε να διαχωριστεί το ποσό σε δύο μέρη. Η Κομισιόν διατήρησε 9 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο των 18 το 50% μέχρι ότου επιτευχθεί υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης. Επιπλέον, με σκοπό να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, εισήχθη ένας νέος μηχανισμός, ο CAS, ως προσωρινό μέτρο. Ο μηχανισμός αυτός θα αρχιθεθεί σε λειτουργία κατά το πρώτο εξάμεινο του 2011. Η δημιουργία του νέου αυτού ειδικού λογαριασμού θα συνεισφέρει στην εγγύηση στο να εγγυηθεί ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν κατευθείαν στην στήριξη του κλάδου, το οποίο και επιθυμούμε. Το νέο πρωτόκολλο μετά την 1η Αυγούστου του 2012 θα λάβει υπόψη, υπόψη του την επερχόμενη αναμόρφωση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής η εντολή αναδιαπραγμάτευσης περιλαμβάνει και μια ρήτρα για πρώτη φορά δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα θα εγκρίνει την εντολή αυτή. Τώρα όσον αφορά την ε, καταπολέμηση της αηλίας IUU, μετά την θέσπιση του κανονισμού η κομισιόν έχει συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές της μαυριτανίας. προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την καλή εφαρμογή των μέτρων αυτών. Τέλος, οι επενδύσεις του αλληλευτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται με βάση το πρόγραμμα δράσης Μαυριτανίας, το οποίο στοχεύει να διευκολύνει την εγκατάσταση ευρωπαϊκών ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεικτών επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών, ε, Μαυριτανικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να εξασφαλίσει τις καταλληλότερες μορφές ΣΔΙΤ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Κάντεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με βάση τη συνδίκη της Λισαβόνας το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ε, τη συμφωνή γνώμη τους, τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα πρέπει ανα πάσα στιγμή να είναι ενήμερο για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Η Πρέπει το 31 Δεκάτου του 2012 να ανανεωθεί Συμφωνία ελευθερική Σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαυρετανίας. Και εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη χρηματοπιστωτική εισφορά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με τα αλλιεύματα. Είναι η μοναδική συμφωνία που επιτρέπει ε, να, ε, γίνονται, να γίνεται αλλία κεφαλοπόδων και οστρακοειδών όπως και με τη Γιουνέα Μπισάου η έλλειψη υποδομής ε, ε, στα λιμάνια είναι υπαρκτή και άρα πρέπει να γίνουν επενδύσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια ευρωπαϊκά σκάφη ε, εμποδίστηκαν από τις μαυρετανικές αρχές χωρίς δικαιολογία. η δουλειά, το έργο των εφοπλιστών δυσκολεύεται λόγω διαφόρων πράξεων της μαυρετανικής πλευράς. Πρέπει να ξεκαθαριστούν τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται για τους Ευρωπαίους εφοπλιστές, οι οποίοι υφίστανται διακρίσεις σχέση με άλλους τόλους που αλλιεύουν στην περιοχή. Θα ήθελα τελικά να μην υποτιμάμε τον κινέζικο παράγοντα σε σχέση με την αλία στη Μαυριτανία που ασκεί μέσω κοινοπραξιών και με την κάλυψη της ε, ε, μαυριτανικής σημαίας επηρεάζει την αλία η οποία πρέπει να υφίσταται κάθε ε, έλεγχο υγειονομικό και εμπορικό και να μην ξεχνάμε την εξάντληση των αλλιευτικών πόρων. Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της αλληλείας γιατί πρέπει να διευκολύνονται οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές. Θα πρέπει η Επιτροπή Αλίας να ασχοληθεί εκ των υστέρων και εκτενώς με την ε, μελέτη Επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε, στο Στρασβούργο είμαστε πολύ καλά όπου έχει ακριβώς την θέση που του αρμόζει αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. That. Το πιασα αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Um, ο κύριος Άσενης έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επιτρόπε Δαμανάκη, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρωτοβουλία των σοσιαλιστών ε, για το ψήφισμα για τη Μαυριτανία έχει ακριβώς να καλύψει ένα κενό μετά τη συνθήκη Λισαβόνας ε, έχουμε έναν πιο ξεκάθαρο ρόλο του Κοινοβουλίου, ένα ρόλο συναπόφασης στα ευρωπαϊκά θέματα. Ε, το Κοινοβούλιο καλείται να επικυρώσει ε, συμφωνίες και διεθνείς αλληλευτικές συμφωνίες και όμως ο ρόλος αυτός του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμα δεν έχουμε έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση, έγκαιρη συμμετοχή για και πλήρη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και αν δεν έχουμε, ε, δεν, οι συμφωνίες αυτές δεν μας έρχονται πριν αρχίσει η εφαρμογή τους. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της Επιτρόπου που αναγνωρίζουμε, ε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το Κοινοβούλιο καλείται να επικυρώσει συμφωνίες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ήδη και ένα χρόνο. Ε, το Κοινοβούλιο δεν πληροφορείται για την πορεία των διαπραγματεύσεων με επίσημο τρόπο και το Κοινοβούλιο προσφάτως έχει δυσκολίες ε, ε, να έχει πρόσβαση σε κείμενα που είναι η εκτίμηση των ε, επιπτώσεων και της πορείας και της εφαρμογής προηγούμενων συμφωνιών. Χρειάζεται να αλλάξουμε πάρα πολλά στις ελευτικές μας συμφωνίες. Πρέπει να αλλιεύουμε εκεί πέρα που υπάρχει πλεόνασμα αλλιευμάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούμε την αρχή της προφύλαξης. Πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την παράνομη και αναρχιαλία πρέπει πραγματικά οι συμφωνίες να έχουν και αναπτυξιακά ωφέλη για τις χώρες με τις οποίες τις, ε, ε, που συμφωνία. Ειδικά για τη Μαυριτανία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και από παράνομη ε, αλία και από χρήση, καταχρηστική χρήση εργαλείων και πραγματικά ο ρόλος και η παρέμβαση του Κοινοβουλίου θα είναι προκειμένου και καλύτερες συμφωνίες και στην περίπτωση της Μαυριτανίας και γενικότερα να επιτευχθούν και να εφαρμοστούν αυτές σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Jag hörde till dem som hade förmånen att besöka i slutet av Εγώ πέρσι ήμουνα στη Μαυριτανία για να αξιολογήσω λίγο η κατάσταση, να δω πώς λειτουργούσε η συμφωνία και είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι μπορώ απέχει η κατάσταση από την επιθυμητή. Διαθέτουμε 25 εκατομμύρια ευρώ στη συμφωνία αυτή και λέμε ότι αυτό είναι το 30% περίπου του ΑΕΠ της Μαυριτανίας. Επομένως αυτό το ποσό δεν είναι μόνο σημαντικό για αυτούς αλλά και για μας. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην ατζέντα του 2020 και λέει πώς πρέπει να βελτιώσει ε, την αξία των συμφωνιών της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, πράγματι αλλάζει η ζήτηση συνεχώς αλλά διερωτώ με πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια που διαθέτουμε. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε δε ότι η συμφωνία λέει ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε και την τοπική αλία. Η ερασιτεχνική αλία όμως ήταν ελάχιστη και ε, αυτό είναι ανησυχητικό διότι επενδύουμε τεράστια ποσά. Θα πρέπει λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, να αλλάξουν τα πράγματα. Θα πρέπει να ε, δούμε τι ακριβώς κάνουμε και με το βλέμμα στο μέλλον έχουμε ευθύνη για τα θέματα αυτά, διότι συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία λήψη απόφαση πλέον βάσει της νέας συνθήκη. και γι' αυτό και υποχρεώμεθα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και για το μέλλον, διότι ό,τι κάνουμε εμείς και ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βασίζεται και στις πληροφορίες που θα λαμβάνουμε. Thank Σας ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ευπρόσδεκτες οι προθέσεις ε, στο, της Κομισιόν στο σχέδιο των κατευθυντριών γραμμών το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ελέγχου των δημοκρατικών αρχών είναι εξαιρετικό. Η ενίσχυση του διαλόγου για να ενισχυθεί η υπεύθυνη αλληλεία είναι και αυτή ιδιαίτερος ε, ευπρόσδεκτη, διότι στις υφιστάμενες συμφωνίες σχεδόν ποτέ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα όσον αφορά ε, πρόσβαση των ευρωπαϊκών σκαφών σε κάποια μόνο είδη ε, αλλιευμάτων. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί οι οι τράτες ανταγωνίζονται τις ε, τράτες της Μαυριτανίας. Ελπίζω ότι αυτό θα περιοριστεί. Τώρα όσον αφορά τα αποθέματα. Η ομάδα ε, ε, μικρής πελαγικής αλίας του 2010 κατέληξε ότι υπήρχε είτε πλήρης είτε υπερεκμετάλλευση κάποιων ε, αλλιευμάτων. Για να είμαι σύντομη, ποιο πλεόνασμα αλλιευμάτων αναμένει η Κομισιόν να βρει στη Μαυριτανία και περιμένει ότι θα στηρίζει τον κλάδο στη Μαυριτανία ακόμα και αν οι ε, δυνατότητες περιοριστούν. Δεν μπορούμε να υπεραλλιεύουμε αυτά τα νερά, να πηγαίνουμε, να παίρνουμε ό,τι υπάρχει και να φεύγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερέρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουν περάσει πάνω από δύο δεκαετίες από το πόση η Κομισιόνα έχει συμφωνίες με την Μαυριτανία και στο παρελθόν σχετίζονται και με το θέμα της συνεργασίας για την διατήρηση του περιβάλλοντος. Το θέμα που τίθεται σήμερα είναι ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής. Γιατί ο τομέας της Αιλίας στη Μαυριτανία έχει πάρα πολύ ελληματική εξέλιξη. Η εξέλιξη της ε, τοπικής ε, παράλληλες αλίας, ε, όλη η βιομηχανία αλίας, ε, η υποδομή, όλα τα σχέδια όσον αφορά την ε, υδατοκαλλιέργεια κλπ. Όλα αυτά ήταν στόχοι που είτε παρέμειναν νεκρό γράμμα, είτε προχώρησαμε πολύ μη μικρά βήματάκια. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετεβάζουν τεράστια κονδύλια για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις, ε, ε, τους φυσικούς πόρους ε, του, της χώρας αυτής εις βάρος των πιο φτωχών που θα έπρεπε μόνοι να τους εκμεταλλευτούν. Χάνει η Μαυρετανία και όσον αφορά και την εκμετάλλευση, όσον αφορά την, το κύκλο εργασιών, όσον αφορά την εξέλιξη. Είναι απαράδεκτο χιλιόμετρα από τις ακτές ε, της χώρας αυτής ε, γίνεται μια βιομηχανική αλία και τα αποτελέσματα είναι ότι τα λεύματα αυτά προσάγονται σε άλλες λιμένες, άλλες λιμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να φροντίσουμε να, να εμπλέξουμε τις αρχές της Μεροτονίας για να έχουμε καλή και σωστή εξέλιξη. Ευχαριστώ κύριε Πετράνευση. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ελευτική Συμφωνία με τρίτες χώρες θα πρέπει να προσφέρει ισορροπία μεταξύ των δικών μας συμφερόντων και της πρόθεσης της ε, βιώσιμης αλίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε ε, σε αυτές τις χώρες τις καλές πρακτικές που εφαρμόσουμε στις δικές μας χώρες. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ισορροπία των συστημάτων. Η συμφωνία ε, με τη Μαυριτανία είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης μείωση φτώχεια, ανάπτυξη δομών για τον τομέα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να προωθεί η βιώσιμη αλεία και ταυτόχρονα να ε, απαγορευτεί η παράνομη αλεία. Ε, δεν αρκεί εάν τα κοινοτικά αλευτικά σκάφη ακολουθούν ε, τις αρχές της βιώσιμης ηλίας. Θα πρέπει όλα τα σκάφη που συμμετέχουν στη συμφωνία αυτή να τηρούν αυτούς τους όρους. Η Μαυριτανία απαιτεί με, στις τρίτες χώρες που συνάπτουν ε, ε αλευτικές συμφωνίες να τηρούν τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα δικά μας σκάφη. Αλλιώς υπάρχει στρέβλωση του αναγνωρισμού και δεν γίνεται η βιώσιμη διατήρηση των φυσικών θερασίων. πόρων. Ευχαριστώ και σας μιλάνε ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κατά την άποψή μου έχουμε δύο προβλήματα. Ένα μεθοδολογικό και ένα ουσία σε αυτή την υπόθεση. Ως προς τη μέθοδο θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φράγα. Χρησιμοποιούμε μια προφορική ερώτηση για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο μετά από τη συνθήκη τη Λεβόνας θα πρέπει να είναι αναφόρετο δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι αυτή η πρακτική θα πρέπει να λάβει κάποια στιγμή τέλο. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε στρατηγική για να παρακολουθήσουμε μια διαδικασία συναπόφεση η διαδικασία θα πρέπει να τηρείται στι φάσει στι οποίε οριμάζει. Εμεί σήμερα θα κάνουμε τη συζήτηση, θα τελειώσει η συμφωνία και εμεί θα πρέπει να πούμε ναι στο τέλο. Αυτή η μεθοδολογία πρέπει να σταματήσει να ακολουθείτε. Ω προ την ουσία, θα ήθελα να επισημάνω μόνον, γιατί συμφωνώ με τα περισσότερα από τα όπω είναι οι συνάδελφοι, ότι θα πρέπει οι συμφωνίε αλεία να μην είναι μόνο εμπορικέ συμφωνίε με τι οποίε αγοράζουμε κεφαλόπεδα με ένα ευρώ το κιλό στη Μαυριτανία. Θα πρέπει να μπορούν να προσμετρήσουν και τη βιωσιμότητα αλλά και τις επιπτώσεις για την οικονομία της συγκεκριμένης χώρας. Να καταλάβουμε πώς είναι οι απασχολούμενοι που αλλάζουν. Αν υπάρχει ποσοστό καινοτομία για την ερασιτεχνική αλεία, να καταλάβουμε πού χρησιμοποιούνται αυτοί οι πόροι και να μην είναι μια απλή εμπορική συμφωνία, αλλά μια συμφωνία αλεία με όλα όσα επισέρχονται εντό αυτή. Ευχαριστώ η κυρία Ανδρέα Παρέα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σε ένα χρόνο εκπνέει η συμφωνία με τη Μαυριτανία και προετοιμάζομαστε για τη νέα συμφωνία. Θεωρώ ότι η συμφωνία με τη Μαυριτανία είναι ένα καλό μέσο, είναι ένα μέσο ανάπτυξης για τη χώρα, αλλά και για τις τομεακές πολιτικές αλληλείας της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι είναι το 29% του ΑΕΠ και είναι η μόνη δυνατότητα ανάπτυξης που έχει η χώρα αυτή. Ενισχύει τη διμερή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαυρετανίας και θα πρέπει να διασφαλίζει και τη βιώσιμη αλληλεία. Μιλάμε για παράνομη αλληλεία και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε και την Επιστημονική Επιτροπή για να προσφέρει και περισσότερα μέτρα ώστε να γνωρίζουν και τι πρέπει να αλλιεύουν ώστε να έχουμε βιώσιμη αλληλεία. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε και τι δυνατότητε των σκαφών. Η επίτροπο αναφέρθηκε και στην αδυναμία τη κυβέρνηση τη Μαυριτανία, η οποία θα πρέπει να αναπτύξει τι διοικητικέ τη δομέ προκειμένου να μπορέσει να προσαμιώσει τι ε, μεθόδους της με τι μεθόδου Ευρωπαϊκής Ένωση και να υπάρχει αντιστάθμισμα για τα όσα ε, προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομική πλευρά. Επίση, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, ζητούμε από την Μαυριτανία να συμπεριλάβει τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προάγει τον εκδημοκρατισμό τη χώρα. Οι αλληλευτικέ συμφωνίε είναι ένα μέσο για να εκδημοκρατιστούν οι χώρε αυτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριο Σάντσε Πρεσέδο, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ζήτησε εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει για τη νέα αλληλευτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαυριτανίας, η οποία θα αντικαταστήσει την ε, ε, υφιστάμενη από 31 Ιουλίου του 2012. Θα πρέπει η συμφωνία να συζητηθεί με ένα πραγματικό πνεύμα συνεργασίας λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βασίζονται στις συνθήκες Λισαβόνας. Θα πρέπει να υπάρχει και ένας βιώσιμος ορίζοντας ε, για τον κοινοτικό στόλο στα ύδατα της Μαυριτανίας. Θα πρέπει να υπάρχει και ίση συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιμη ανάπτυξη του αλλιευτικού τομέα της Μαυριτανίας που θα πηγαίνει πέραν του οικονομικού τομέα και θα πρέπει να ενισχύσει και το διεθνέ δίκαιο και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. το ποσό που διαθέτουμε στην πραγματικότητα είναι το 1 τρίτο του προπολογισμού τη Μαυριτανία. Και αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί σωστά, να προάγει την ε, βιώσιμη αλληλεία και να βοηθά τον τομέα και να σε επιτρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλληλεία ενισχύοντας τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που υπάρχουν ε, επί του παρόντος. Ευχαριστώ πολύ. Στη διαδικασία κάτσι διάει ο κύριος Βαρέντσα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για την παρουσίασή τη. Ο ελεκτικό στόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετό καιρό στα μαυριτανικά ύδατα και λόγω του μακρού αυτοχρονικού διαθήματο έχουμε πολύ καλέ και ιδιαίτερε σχέσει με τη Μαυριτανία. Αυτό σημαίνει ότι έτσι μπορούμε να εμπλακούμε στην Αφρική για να βοηθήσουμε να πλησιάσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την Ελληνία εταιρική σχέση όσον αφορά την αλληλεία, εντό για τα πελαγικά είδη, είναι στρατηγική σημασία όχι μόνο για την επιβίωση των ελευτικών μα στόλων, αλλά είναι σημαντική και για την επιστημονική βιομηχανία. Πρόκειται για συμφωνίε που είναι προ όφελο και των δύο πλευρών και έχει κάθε συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει αυτέ τι συμφωνίε. Ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσουμε οι διαδικασίε να είναι διαφανεί. Και αυτό είναι χρήσιμο για όλους τους ενδιαφερομένους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μόλτσερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν εξετάζουμε την αδευτική Συμφωνία με την Βρετανία, ξέρουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για μια συμφωνία σε πολύ ευαίσθητο χώρο. Ένας χώρος ο οποίος Βλέπουμε όπως η Βόρεια Αφρική αυτή τη στιγμή πώς βρίσκει το επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Θα πρέπει βέβαια η συμφωνία αυτή να είναι προ όφελο στο οικονομικό των ενδιαφερομένων, αλλά θα πρέπει να ακολουθούμε και οικολογικά κριτήρια. Εάν η συμφωνία αυτή αποτελεί το 1 τρίτο του προπολογισμού της Μαυρετανίας, καταλαβαίνουμε τη σημασία της. Από την άλλη μεριά, ο ελευτικός στόλο στόλος της Ένωση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός οικονομικός ε, το ένα είναι το θέμα το οικολογικό, το άλλο είναι ότι θα πρέπει με μια τέτοια συμφωνία να ενδυναμώσουμε τον εκδοκιμασμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια χώρα που ενδεχομένω θα έχει τα ίδια προβλήματα όπω και άλλε χώρε τη Βορειοαφρικής. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την κατάσταση και ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστώ η κυρία Δαμανάκη. like thank... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που παρενέβησαν και να πω ξεκάθαρα ότι χαιρετίζω όλους ιδιαιτέρως την συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις και αυτής της συμφωνίας και των άλλων συμφωνιών. Θα ήθελα, θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μια νέα συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Εκτελεστικής Επιτροπής και Κοινοβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτής της συμμετοχή τους και θα πρέπει να, συμφων... να σεβαστούμε αυτή τη συμφωνία. Στα πλαίσια της συμφωνίας πλαίσιο είμαι εδώ για να διευκολύνω την συμμετοχή σας και την ενημέρωσή σας. Και προτίθεμαι να συνεργαστώ για οτιδήποτε μπορούμε να βελτιώσουμε. Αυτό επί της μεθόδου και διαδικασίας. Όσον αφορά την ουσία, χρειαζόμαστε προσεκτικό και ε, ισορροπημένο τρόπο προσέγγισης λόγω της μεγάλης σημασίας της χώρας αυτής και λόγω του, των εξελίξεων που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στον λόγο γεωγραφικό τομέα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης των πλεονεσμάτων και γενικά των πρώτων υλών και από την άλλη μεριά των συμφερόντων του στόλου μας για να διευκολύνουμε το στόλο αυτό να πάει εκεί και να μπορέσει να παίξει σε ένα ίσο πεδίο παιδής. Δεν είναι τα μόνα σκάφη που βρίσκουν εκεί, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες στην περιοχή και θα πρέπει να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε να είναι ίση η όρη για όλους. Θα πρέπει να διατηρήσουμε και μια άλλη ισορροπία. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα χρήματα που δίνουμε να φτάνουν στα χέρια των πραγματικά ε, ενδιαφερμένων. Ε, πρέπει να βελτιώσουμε όλες τις διαδικασίες όπου το χρειάζεται η χώρα αυτή. Είναι πολύ λεπτό το θέμα λοιπόν. Και ταυτόχρονα μπορώ να συμφωνήσω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα επιστημονικά στοιχεία και περισσότερες συγκεκριμένες, συγκεκριμένες συμβουλές και στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα την κατάσταση εκεί. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι την επόμενη εβδομάδα να στραφούμε στο Συμβούλιο και να μπορέσουμε να έχουμε μια πρώτη εντολή για αυτές τις διαπραγματεύσεις και κατόπιν θα ενημερώσουμε συγκεκριμένα και μόνιμα την Επιτροπή Αλίας του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρώτη των διαπραγματεύσεων. Ε, τελευταία αναλύση έχω να σας πω ότι αν νομίζετε ότι αυτή η συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε πραγματικά όλοι θα κερδίσουν από μια τέτοια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, Επιτρόπε. Ευχαριστώ όλου που συμμετείχαν στην συνεδρίαση. Η ψηφοφορία θα εξελιχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου. Το επόμενο θέμα σήμερα συνέντευξη είναι η προβολική ερώτηση προ την Εκτελεστική Επιτροπή όσον αφορά τη στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού.